Να ξεκινήσουμε τις ε, ψηφοφορίες. Έχω δύο ανακοινώσεις να κάνω και θα ήθελα την προσοχή σας. Η πρώτη ανακοίνωση αφορά τον σεισμό στην Ταϊβάν. Στην έναρξη της ε, συνεδρίασης σκεφτόμαστε τα θύματα του ισχυρού σεισμού στην Ταϊβάν χτες, ε, κάποια τα οποία ακόμα αγνοούνται. Ευχόμαστε στις ε, οικογένειές τους και στα σωστικά συνεργεία που ακόμα εργάζονται καλή δύναμη. Η δεύτερη ανακοίνωση. η